Η ημερήσια διάταξη είναι μία προφορική ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ ιδίω σε ό,τι αφορά τη δίωξη των φερόμενων ως ομοφιλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία. Πρώτα θα δώσω τον λόγο στους πέντε συντάκτες της προφορικής ερώτησης και πρωτίστως την κυρία Σοράγια Πώς. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από το Φεβρουάριο λαμβάνομαι τρομακτικές αναφορές από την επαρχία της Τσετσενίας ε, αποτρόπες πράξεις ε, σε βάρος ομοφιλόφιλων. Οι κυβερνητικοί λειτουργοί λέγουν ότι δεν υπάρχουν ομοφιλόφιλοι στην Τσετσενία. Παράλληλα όμως ε, οι πραγματικοί ομοφιλόφιλοι, φερόμενοι ως ομοφιλόφιλοι ε, ε, βασανίζονται και οι φίλοι τους πληρώνουν τεράστια ποσά για να τους απελευθερώσουν από τις φυλακές καμπάνια κατά των ομοφιλόφιλων ε, επηρέασε τα δικαιώματα πολλών οικογενειών. Ε, πολλές φορές ε, οι οικογένειες δολοφόνησαν τα παιδιά τους γιατί ντρέπονταν που ήταν ομοφιλόφιλα. Αυτά συμβαίνουν όταν η πολιτική ε, δρά όσοι αν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για λίγους και ε, ε, ακολουθούν απάνθρωπες πολιτικές. Ε, η προσπάθεια είναι η ισότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό έχουμε ιδιαίτερο καθήκον να προστατεύσουμε ε, τα πρόσωπα ΛΟΑΔΜ που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Η βάση για την ε, ερώτηση είναι πώς θα διασφαλιστεί ο σεβασμός των κατευθυντηρίων γραμμών για τους ΛΟΑΔΜ. Ε, πέντε ακτιβιτές ε, κρατήθηκαν στη Μόσχα όταν ζήτησαν έρευνα ε, για τα εγκλήματα στην Τζετζενία. Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν. σήμερα θα πρέπει να βοηθήσουμε την κοινότητα των ΛΟΑΔΜ στην Τσετσενία της Ρωσίας. Uh, uh, Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Α, η κυρία Ουλρίκε Λούνατσεκ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αύριο είναι η Διεθνή ημέρα καταπολέμησης της ομοφοβίας και γι' αυτό φορά αυτό το αεροαράνιο τόξο εδώ για να υπενθυμίσω σε όλους όσοι μας ακούν και μας βλέπουν ότι είναι μια μέρα που θα πρέπει όλοι να υψώσουμε το ανάστημά μας, όπως το κάνουμε εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εναντίον της ομοφιλοφοβίας, εναντίον όλων των ειδών βίας που πλήττει βία όλους τους ανθρώπους στην Ευρώπη και στις άλλες υπήρους. Και γι' αυτό λοιπόν η συζήτηση αυτή είναι ειδικά αφιερωμένη στις αναφορές που για τα τεκτενόμενα στην Τσετσενία τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχουν αναφορές για βασανιστήρια εκατοντάδων ε, ανδρών που είναι γκέι, που θεωρούνται γκέι και τρεις από αυτούς ε, τουλάχιστον έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους και τους ζητείτε με τα βασανιστήρια να αποκαλύψουν την ταυτότητα και άλλων ανθρώπων. Είναι μια ζωή μέσα στο φόβο και κανείς αυτό το πλανήτη δεν πρέπει να τη ζει αυτή τη ζωή και κανείς ε, από αυτούς που προστατεύουν ε, τους ε, ενόχους δεν πρέπει να μείνει μακριά από τη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να αποδώσει λογαριασμό και χαίρομαι διότι υπάρχει ευρία στήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες σχεδόν. Ζητούμε από τη Ρωσική Ομοσπονδία, από το καθεστώς της Τσετσενίας να προστατεύσει τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΑ και να υψώσουν το ανάστημά τους όλοι. Να πούμε ότι όλα αυτά είναι ε, απολύτως προστατευόμενα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάτι που υπήρχε πάντοτε από απαρχής της ανθρωπότητας σε όλες τις κοινότητες, σε όλους τους λαούς, σε όλους τους πολιτισμούς και πρέπει να δοθούν σωστές κατευθυντήριες γραμμές. Να μεριμνήσουμε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές μας εφαρμόζονται παντού στο πλανήτη μας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΜ και οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες να πράξουν τα δέοντα. Χαίρομαι και εκτιμώ ιδιαιτέρως διότι υπάρχει σχετική δράση ε, στα χρώματα του ουράνιου τόξου θα φωτιστεί το κτίριο της υπηρεσίας της οποίας προείσταται ο Επίτροπος κ. Στυλιανίδης ε, ως πάλι μια συμβολική δράση υπέρ των δικαιωμάτων ε, του ατόμου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μαρίν Μπιόρκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, πολύ δυσκολεύτηκα να διαβάσουν αυτή την έκθεση για τους φόνους και για τις απειλές που υφίστανται οι ομοφυλόφιλοι. Είναι ε, φρικτές οι διώξεις και είναι δύσκολο κανείς να τις ε, ε, καταπιεί, αν θέλετε, να τις χωνέψει. Είναι ακραία βία αυτή που παρουσιάζεται στην έκθεση και ευτυχώς είναι κάτι που συμβαίνει εξαιρετικά ε, σπάνια. Ωστόσο, είναι κάτι που σκοτώνει ανθρώπους εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε και το, το περιστατικό στο συμβάν στο κλαμπ Ορλάντο, όπως γνωρίζετε. Ε, υπάρχει μεγάλη καταπίεση και εναντί των νέων και των ενηλίκων στις κοινωνίες μας και στη Τσετσενία αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ε, αυτό στο οποίο μπορούμε να οδηγηθούμε όταν, έχουμε, όταν υπάρχει αυτή η ομοφοβία ε, σε ακραίο βαθμό. Θα πρέπει όλοι να δράσουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση για να μπορέσουν να διερευνήσουν τι ακριβώς συνέβη και οι υπόλογοι θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε να συμβαστούμε με τίποτα λιγότερο. Από εκεί και πέρα Υποτίθεται ότι στην οικογένεια του πρέπει κανείς να νιώθει ασφαλής και στα χέρια της αστυνομίας. Και όμως οι οικογένειες και η αστυνομία είναι αυτές που συνέβαλαν στη δίωξη των ομοφυλοφιλών και στο θάνατό τους τελικά. Η ομοφοβία είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό της πατριαρχικής κοινωνίας, είναι κάτι το απολύτως αποτρόπαιο. Το καταδικάζουμε απερίφραστα και άρα οφείλουμε να δράσουμε εναντίον της ομοφοβίας. Είναι κάτι που πλήττει την Τσετσενία αλλά και τις δικές μας χώρες. Έχουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε ε, αν ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις κοινωνίες μας σε συνθήκες ε, αξιοπρέπειας και οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πέτρας για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Κύριε Επίτροπε, η βίαιη εκστρατεία εναντίον των ομοφιλοφίλων στην αυταρχική ε, τετσενία του Καντήροφ δείχνει πόσο λίγο ε, υπολογίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτό το τμήμα της Ρωσίας σήμερα η συνεχιζόμενη τρομοκρατία και δίωξη της αντιπολίτευσης αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, των δημοσιογράφων, τώρα περιλαμβάνει και τους ΛΟΑΔΜΑ. Δυστυχώς όλα τα εγκλήματα στην Τσετσενία που έχουν συμβεί δεν είναι μεμονωμένα συμβάντα είναι ένας κοινό παρανομαστής που δείχνει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρωσία στο σύνολό της. Να θυμηθούμε ότι τον μήνα Μάρτιο η Ρωσία υιοθέτησε μια οπισθοδρομική νομοθεσία η οποία αποποινικοποιεί την οικιακή βία. Και τώρα έχουμε την ιστορία με τους ΛΟΑΔΜΕΣ. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι βέβαιη ότι η πολιτική μας απέναντι στη Ρωσία περιλαμβάνει και το θέμα των εγκλημάτων εις βάρος των ΛΟΑΔΜ στην Τσετσενία. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση αυτή. Η ομοφοβία ανήκει στο φρικτό παρελθόν μας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής και συνεισηγητής είναι ο κύριος Ντέμερς Μέκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αύριο 17 Μαΐου στη χώρα μου θα κυματίζουν στη Φλάνδρα οι σημαίες του ουράνιου τόξου και στο Δημοτικό Μέγαρο και ε, γενικά στο Κοινοβούλιο το Φλαμανδικό ε, γιατί δείχνουμε ότι έγιναν αγώνες και προσπάθειες ε, για ε, το σεβασμό των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜΑ. Δυστυχώς τα προβλήματα παραμένουν σε πολλές χώρες και η κατάσταση στην Τσετσενία είναι πραγματικά τρομακτική. Συνεχίζει ο χειμώνας δυστυχώς στην περιοχή αυτή του Καυκάσου λέει ο ομιλητής και εκατοντάδες άνθρωποι είναι φυλακισμένοι διότι υποτίθεται ότι είναι ομοφιλόφιλοι. Οι ενέργειες του Προέδρου Νακαντήροφ ε, για να δείξει ότι δεν υπάρχουν ομοφιλόφιλοι στην χώρα του αποδεικνύουν ε, αν θέλετε την ε, έλλειψη καλής θέλησης του καθεστώτος αυτού. Και φυσικά ε, το Κρεμλίνο υποστηρίζει το καθεστώς ε, του Γκρόσνη και επιτίθεται συστηματικά και στη Μόσχα σε αυτούς που διεκδικούν τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΑ. Και το Συμβούλιο της Ευρώπης στην τελευταία του έκθεση είπε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει καταφέρει τίποτα ε, για να βελτιώσει την απαράδεκτη κατάσταση η οποία σοβεί στην Τσετσενία. Πρέπει να υπάρξει μια ανεξάρτητη έρευνα, αλλά κανένας βέβαια δεν περιμένει από τη Ρωσία να το κάνει αυτό. Το θέμα είναι λοιπόν τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εφαρμοστούν οι κανόνες που ισχύουν και για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα και ειδικότερα και για τους ΛΟΑΔΜΑ. Θα πρέπει επιτέλους οι ρωσικές αρχές να σεβαστούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Ε, Ευχαριστώ. Και τώρα ε, για την ε, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Επίτροπος Χρήστος Τηλιανίδης έχει το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Διακρίσεις και επιθέσεις δεν πρέπει να γίνονται σε βάρος κανενός. Αυτή η αρχή έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της αντίληψής μας για την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ε, πρόκειται για μια ευρωπαϊκή αρχή προφανώς και πιστεύομαι ότι η αξία αυτή πρέπει να είναι καθολική. Θυμίζω ότι το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για να προωθήσει ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ΛΟΑΔΜ. Οι διπλωματικές προσπάθειες της Ένωσης σε αυτό το τομέα περιστρέφονται γύρω από τέσσερις προτεραιότητες. Πρώτον, κατάργηση των διακριτικών πολιτικών και νομοθεσιών και, και ε, την ποινικοποίηση, προώθηση ισότητας και μη διακρίσεις στον τόπο εργασίας, στην υγεία και την εκπαίδευση, ε, καταπολέμηση της ε, ατομικής βίας σε βάρος των ΛΟΑΔΜ και τέλος ε, υποστήριξη των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανάλογα με την περίσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δρά με ήπια διπλωματία, δημόσιες ε, δηλώσεις και παρουσίαση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ στις συζητήσεις με τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει και την κοινωνία των πολιτών που είναι το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σήμερα, όπως είπατε εσείς οι συντάκτες, ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε κάποιους πολύ σοβαρούς υπενιγμούς σε βάρος ομοφιλοφίλων ανδρών στη Τσετσενία. Η δίωξη των ομοφιλοφίλων που οδηγεί σε βασανισμό, ε, δολοφονίες, απαγωγές είναι ορισμένες πολύ ανησυχητικές εξελίξεις στη Τσετσενία. Οι αρχές της Τσετσενίας ε, εμέσως δικαιολογούν τη βία και οι ρωσικές ε, ομοσπονδιακές αρχές υποβαθμίζουν το θέμα και θεωρούν ότι οι αναφορές αυτές είναι fake news και υπερβολές. Δυστυχώς μέχρι τώρα οι ρωσικές αρχές δεν ανέλαβαν αποτελεσματική δράση για να τεθεί τέλος στη βία και να προστατευθούν τα θύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κράτη-μέλη της και άλλες χώρες ε, που πιστεύουν τα ίδια πράγματα όπως και οι οργανώσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν τις ε, ομότητες σε βάρος των ομοφιλοφίλων και δεκάσονται υπέρ μιας πλήρους έρευνας που θα φωτίσει το τι συνέβη. Μόλις χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης συζήτησαν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων το θέμα για να αξιολογήσουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο να βοηθηθούν τα θύματα ε, αυτών των καταχρήσεων. Βέβαια, η είπατε εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνη ε, έθεσε τις σοβαρές μας ανησυχίες άμεσα στον Υπουργό Λαυρόφ όταν τον είδε στις 24 Απριλίου στη Μόσχα. Ετώνησε την ανάγκη να τέθει άμεσα τέλος στις διώξεις κατά των ομοφιλοφιλών στην ε, Τσετσενία και να, ερευνηθεί, να ερευνηθούν αυτές οι αποτρόπες εκθέσεις. Δυστυχώς η απάντηση του Υπουργού Λαυρόφ αργότερα που αργότερα επανελήφθησαν στην ε, συνέντευξη τύπου είναι ότι οι ρωσικές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν αποδείξεις ότι οι διώξεις ε, όντως συνέβησαν. Ενώ στη Μόσχα είπα ότι εκπρόσωπος είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφων, είναι ανησυχητικό ότι οι δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν την εκστρατεία βίας ε, με τη σειρά τους έγιναν στόχος άμεσων απειλών από την ηγεσία της Τσετσενίας και αναγκάστηκαν να φύγουν από την Τσετσενία, να διαφύγουν. Αυτή είναι η κατάσταση επιτόπου. Ζητήσαμε από τους πρέσβεις στη Μόσχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουν τους άνδρες που αποτέλεσαν στόχο καταχρηστικών πρακτικών, ιδιαίτερα εκείνων που ακόμα φοβούνται για την ασφάλεια τους και την προστασία τους. Κάποια κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να βοηθήσουν. Ό,τι κάνουν θα γίνει ήσυχα και χωρίς φανφάρες για να προστατευθούν τα θύματα. Εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσουμε να ζητούμε από τις ρωσικές αρχές για μια πλήρη έρευνα των υποθέσεων των δολοφονιών, απαγωγών και βασανισμών ομοφιλοφίλων ανδρών στην Τσετσενία. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει και όποιος ε, βρεθεί να είναι υπέτειος ε, να πάει στην δικαιοσύνη. Ε, είμαστε πεπισμένοι ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Δίνουμε τώρα ε, το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, 1,5 λεπτό, έχετε το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους και να εκφράσω την αγανάκτησή μου, διότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση για αυτούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί ε, στην ε, Τσετσενία επειδή είναι φερόμενα ΛΟΑΔΜΑ. Ε, αυτό το κυνήγι το συστηματικό των μαγισσών λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού της είναι κάτι το απαράδεκτο τρομακτικό. Δεν μπορούμε να σιωπήσουμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε ενωμένοι και είναι θετικό ότι ο πρόεδρός μας άμεσα αντέδρασε απέναντι στα εγκλήματα αυτά και πρέπει να υπάρξει και περαιτέρω δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να ζητήσουν την απελευθέρωση όλων αυτών που κρατούνται παράνομα και πρέπει να βοηθηθούν τα θύματα. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να διερευνήσει τα εγκλήματα αυτά και να τα καταδικάσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη. Και επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν διώξεις εις βάρος αυτών που καταδικάζουν και καταγγέλουν την βία εις βάρος των ΛΟΑΔΜΑ. Ε, οι υποχρεώσεις μας ε, απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη δεν επιτρέπουν διακρίσεις ε, ανάμεσα στους πολίτες λόγω της διαφοράς τους ή λόγω της φερόμενης διαφοράς τους. Σήμερα το μίσος, η ομοφοβία και ο φόβος της διαφορετικότητας δεν θα πρέπει παρά να καταδικάζονται. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ θα υποστηρίξω το ψήφισμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής ε, Ομάδας η κυρία Βαλενθιάνου. Ήθελες να μείνεις ανέστητος για να σε αφήσουν ήσυχο, αλλά σου έκαναν ηλεκτροσόκ για 20-30 δευτερόλεπτα. Λιποθυμούσες και σε ξαναξυπνούσαν. Αυτό Αυτά είναι μαρτυρίες ενός νεαρού Τσετσένου που κατάφερε να ξεφύγει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που υπάρχουν στη Τσετσενία και σε, αυτή τη, και σε αυτό το μέρος και σε άλλα μέρη του κόσμου το να έχει συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό μπορεί να σε οδηγήσει στο θάνατο ή στο να ζήσει υποκαθεστώς τρομοκρατίας και φόβου. Η κυβέρνηση βέβαια μπορεί να λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την ομοφιλοφιλία στη Τσετσενία γιατί στη Τσετσενία τους ή άλλως δεν υπάρχει ομοφιλοφιλία. Είναι μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά το κρεμπλίνο κοιτάζει από την άλλη μεριά. Ωστόσο, η Ρωσία έχει συνυπογράψει τη συνθήκη, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση που απαγορεύει τα βασανιστήρια και τις διακρίσεις για οποιοδήποτε λόγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ουσιαστική δράση για να προασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜΑ. Και θα πρέπει να το πράξουμε αυτό στις σχέσεις μας με τις λοιπές χώρες. Όλα αυτά πρέπει να τα θέσουμε επιτάπητο στη συζήτηση με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε εμείς να κοιτάξουμε από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε στους εαυτούς μας, γιατί όσοι ε, υποφέρουν από αυτές τις διώξεις, το μόνο που έχουν είναι τη δική μας φωνή. Μόνο η δική μας φωνή έμεινε για να τους υπερασπιστεί. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Άλντε, ο κύριος Φέντερλη. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ σαφή της δήλωση. Τονίζετε τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ξεκάθαρα μίλησαν, έστειλαν ένα σαφές μήνυμα. Το ψήφισμα θα τύχει ευρεία στήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για να δείξουμε στη Ρωσία και στη Τσετσενία ότι τέτοιου είδους τάσεις δεν μπορούν να είναι αποδεκτές κυρία Κοράτσα Μπίλτε μίλησε για τους, ε, για τους ανθρώπους που είναι υποκράτηση και που πρέπει βεβαίως να απελευθερωθούν. Όσοι έχουν διωχθεί από τη χώρα θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ξαναενωθούν με τις οικογένειές τους. Αυτή η κάθαρση που έχει γίνει από την έναρξη του Ραμαζανίου ε, πρέπει να σταματήσει. Έγινε λόγος για οι οικογένειες τους οποίους παρακίνησαν να πάρουν τη ζωή των γιών τους που έχουν κάνει αυτές τις επιλογές ή αλλιώς θα ε, αντιμετωπίσουν ολόκληρες οικογένειες τις ε, συνέπειες αυτές. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την πολιτική Πούτιν, η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Τσετσενία είναι ένα εργαστήριο για αυτόν. Εκεί εφαρμόζει την αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θέλει να επιφυλάξει και στους υπόλοιπους. Θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κορνέλια Έρνστ από την ΚΟΕ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρο Καντήροφ λέει ότι δεν υπάρχουν ομοφιλόφιλοι στην ε, Τσεσενία. Αυτό είναι παραμύθι, όπως ότι με τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά εδώ δεν έχουμε μόνο ομοφιλόφιλους, έχουμε τους ΛΟΑΔΜΑ. Αυτό είναι δώρο της ανθρώπινης φύσης που πρέπει να, η διαφορετικότητα πρέπει να την υπερασπιστούμε. Κυνήγι μαγισσών ε, δεν επιτρέπεται. Πρέπει να σταματήσει, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από κυβερνήσεις. Και ε, δεν είναι δυνατόν να ε, συλλαμβάνονται και να δολοφονούνται οι ομοφυλόφιλοι στην Τετζενία. Και το κράτος που παρακολουθεί χωρίς να κάνει τίποτα είναι εξίσου συνένοχο πρέπει να απελευθερωθούν όσοι συνελήφθησαν για τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ε, οι καταναγκαστικές επεμβάσεις, ο καταναγκασμός ε, καταδικάζεται παντού και στα κράτη-μέλη μας. Και βέβαια είναι σημαντικό να ε, δίνουμε άσυλο στους ανθρώπους αυτούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν διώκονται για αυτούς τους λόγους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Πρασίνων, η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς για ένα λεπτό. Η πρώτη είδηση για το Πογκρόμ που τη διάβασα στο δίκτυο ε, έλεγε ότι τον ε, πέταξαν έξω από την πόρτα και τον απείλησαν ότι θα τον βασανίσουν. Αυτό ήταν μια πρώτη δημοσίευση και μας απασχόλησε, μας συγκλώνησε ε, ως είδηση από τη Τσετσενία. Αυτό είναι καλό, αλλά από την άλλη είμαι και απεσιόδοξη, γιατί πιστεύω αφενός ότι είναι σωστό η Άγγελα Μέρκελ και η Φεντερίκα Μογκερίνη να ε, καταδικάζουν το πογκρόμ αυτό. Είναι καλό ότι ασκήθηκαν πιέσεις στον πρόεδρο Πούτιν, ενδεχομένως θα μπορέσει έτσι να αποτραπεί ένα νέο πογκρόμ, αλλά δεν σταματούμε έτσι τη συστηματική καταπίεση, της διώξει, τη βία σε βάρος των ομοφιλοφίλων και άλλων σεξουαλικών μειονοτήτων στις χώρες αυτές. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται να παρακολουθούμε και να προσέχουμε την κατάσταση. Αλλά αυτό που έκαναν οι σκανδιναβικές χώρες ε, με απλή δυνατότητα εισόδου για ομοφιλόφιλους από την Τσετσενία και διαδικασίες ασύλου, αυτό πρέπει να το προωθήσει τάχιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ομάδας EFDD, η κυρία Μάργκοτ Πάρκερ, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε. Οι αναφορές από την Τσετσενία είναι πάρα πολύ ανησυχητικές. Είναι κατανόητο ότι σε ένα σύγχρονο κράτος πολιτισμένο η ελευθερία, η υγεία κάποιου απειλείται λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού του. Η τσετζενική κυβέρνηση ολισθαίνει στη βαρβαρότητα ε, και πραγματικά ε, συλληπούμε τις οικογένειες των θυμάτων. Η Ρωσία επεκρίθη πολύ ε, σε σχέση με τη στάση τους, στους ομοφυλόφιλους. αλλά τώρα οι Τσετσένοι πάνε σε άλλες ακρότητες. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι όλα αυτά δεν είναι ανεκτά. Θα πρέπει να γίνουν ανακρίσεις, έρευνες και να σταματήσουν οι ε, διώξεις στην Τσετσενία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάρομι Στέτινα, 1,5 λεπτό τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς του καθεστώτος Καντήροφ είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται πλέον να αποδειχθεί. Στην ουσία είναι μια συνέχιση, συνέχεια μάλλον, ε, του, της σταλινικής περίοδου και φυλακίζει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης τις ε, μη υπάκουες ε, μειονότητες. Μετά από την καταστολή από τον ρωσικό στρατό και την προσπάθεια ανεξαρτησίας της Τσετσενίας ε, επικράτησε μια, ένα καθεστώς το οποίο μάλιστα αύριο γιορτάζει την επέτειο της υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στον Γέλτσιν και τον Μασκάροφ το 1997. Ε, η υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τσετσενίας, η κυρία Αμινάτ, είπε ότι ο πόλεμος αυτός εις βάρος της Τσετσενίας δυστυχώς οδήγησε στο θάνατο 100.000 ανθρώπων. Η Ρωσία κατέστρεψε την οικονομία της Τσετσενίας. Ο ρωσικός στρατός με τους συστηματικούς βομβαρδισμούς κατέστρεψε πόλεις ολόκληρες. Ε, φυσικά η Ρωσία ε, παραβίασε όλα τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα, χρησιμοποίησε και χημικά όπλα και η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Αυτά δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παντζέρη έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Την προηγούμενη Πέμπτη απελευθερώθηκε ο Γιούρι Γκουγιάννα, ένας Ιταλός υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχε, ε, είχε συλληφθεί από τις ρωσικές αρχές επειδή είχε διαμαρτυρηθεί ε, στη Μόσχα για την κατάσταση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παραβίαση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜΑ. Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα και όχι μόνο δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους πολίτες, αλλά υποβάλλονται σε βία, σε βασανιστήρια, λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους. Υπάρχει ένα κατασταλτικός μηχανισμός ο οποίος έχει σαν στόχο τον εντοπισμό, την σύλληψη και τον βασανισμό των φερόμενων ως ομοφιλοφίλων. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε το μέγεθος του προβλήματος. Εγώ ε, νομίζω όμως ότι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας ε, δεν ε, ήταν η σωστή. Ο συνομιλητής μας δεν είναι εύκολος συνομιλητής, αλλά θα πρέπει να καταγγείλουμε την κατάσταση αυτή να επιστήσω την προσοχή σας και στις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου. Θεωρώ ότι το έγγραφο μας ζητά κατά συνείδηση να εκφραστούμε ε, για μια ακραία κατάσταση όπως της Τσετσενίας την οποία πρέπει να καταγγείλουμε αλλά και στα σύνορα μέσα, τα σύνορα της Ευρώπης ε, ε, άνθρωποι που ανήκουν στην μειονότητα των ΛΟΑΔΜ την χάνουν καταπίεσης. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Το λόγο θα δώσω τώρα στην κυρία Βίκστρομ. Ένα λεπτό. Είμαστε μάρτυρες τρομερών εγκλημάτων εις βάρος των ομοφιλοφίλων στην όλο και πιο Ισλαμική Τσετσενία την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα νέος 17 ετών ε, αυτοκτόνησε και δολοφονήθηκε επειδή η οικογένειά του δεν ανέχτηκε την ομοφιλοφιλία του. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ενθαρρύνεται έμεσα από το καθεστώς. Υπάρχει εκαθάριση συστηματική με βάση τις προτιμήσεις της ε, σεξουαλικές των πολιτών. Και αυτό φυσικά ε, εις βάρος όλων των ε, ρυθμίσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει εμείς να αντισταθούμε, θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ευάλωτους ανθρώπους, θα πρέπει να πιέσουμε τον κύριο Πούτιν έτσι ώστε να σταματήσουν αυτές οι απαράδεκτες ε, ε, οθήσεις προς ε, φόνους τιμής τις οποίες προωθεί το καθεστώς της Τσετσενίας. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε αυτά τα φρικτά εγκλήματα στην άμεση γειτονία μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φορέντσα έχει το λόγο 1,5 λεπτό. Νομίζω ότι ένα από τα πιο σοβαρά χαρακτηριστικά της υπόθεσης αυτής είναι οι δηλώσεις τις οποίες έκανε η τσετσενική κυβέρνηση για την ανυπαρξία ομοφιλόφιλων στην συγκεκριμένη χώρα. Νομίζω ότι η μόνη και μόνη η συγκεκριμένη δήλωση του Καντήροφ μας οδηγεί στο να αναζητήσουμε την εμβέλεια των διακρίσεων, της καταστολής και των ε, βασανιστήριων ενός, ε, μια κουλτούρας η οποία ε, εδράζεται στην άρνηση αναγνώρισης της ύπαρξης των ΛΟΑΔΜΑ. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο από πλευρά μα όχι μόνο να εκφράσουμε την άποψή μα μέσω τη έγκριση ενός ψηφίσματο αύριο, αλλά να λειτουργήσουμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία δυνατότητα άρνηση ε, πραγματική ή συμβολική των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ. Ευχαριστώ την κυρία Φορέντσα. Η κυρία Χάουταλα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Επίτροπο για την πολύ ισχυρή του παρέμβαση για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όλες τις δυνατότητες που έχει για να καταγγείλει και να καταδικάσει αυτές τις θρικαλαιότητες ε, που ακούμε τους τελευταίους δύο μήνες. Αυτές οι φρικτές διώξεις από τη βία συνδέονται με την έμφαση στην οποία δίνουν σε αυτό το οποίο αποκαλούν αυτοί οι παραδοσιακές αξίες και σύμφωνα με αυτούς, σύμφωνα με τις παραδοσιακές αξίες η ομοφιλοφιλία είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και συνδέεται επίσης και με την αποποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία πρόσφατα γιατί σύμφωνα με τις παραδοσιακές αξίες τα ενίκομοι ενδύμω. Όμως είδαμε βεντέτες να ε, οξύνονται Και στη Τσετσενία σε γενικές γραμμές η κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσχερής, ε, διαπράττονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, καίγονται γραφεία από τις δυνάμεις ασφαλείας, άνθρωποι βασανίζονται, όλα αυτά πρέπει να τα καταδικάσουμε απερίφραστα. Ευχαριστώ πολύ. Τάνια Φαγιών από τους Σοσιαλιστές για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε 10 μέρες θα ξεκινήσει το Ραμαζάνι και για την πλειονότητα των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο είναι μια περίοδος προβληματισμού και ε, ατένισης της ζωής. Ωστόσο είναι ένας μήνας που χαρακτηρίζεται από τρόμο και φόβο για, τους, ε, για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες στη Τσετσενία οι οποίες ε, γιατί στη Τσετσενία έχει τεθεί ο στόχος να εξαλειφθεί ο κοινότητα ΛΟΑΔΜΑ μέχρι την έναρξη του Ραζεμασανίου από τη χώρα αυτή. Αυτά είναι τα φρικτά μηνύματα που φτάνουν στα αυτιά μας από τη χώρα αυτή και οι μαρτυρίες των γκέι που βρίσκονται στα στρατόπεδα κράτησης είναι πραγματικά αποτρόπιες και αδυνατό να διανοηθώ και να φανταστώ τι θα συμβεί αν αποφασίσουν οι αρχές της Τσετσενίας να εφαρμόσουν τις ίδιες μεθόδους και ε, στο γυναικείο λεσβιακό πληθυσμό ή στο πληθυσμό των ατόμων με αναπηρίες. Σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως αυτών τα οποία υποσχέθηκε η Ρωσία δεν έχει κάνει τίποτα και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ανέκαθεν υπήρχαν και οι και πάντοτε υπήρχαν και στη Τσετσενία και θα πρέπει να συνεχίσουν να ε, ζουν ανεμπόδιστα. Οι δηλώσεις του Προέδρου της Τσετσενίας αποτελούν όνειδος, οι δηλώσεις του οι δημόσιες σε διεθνές ε, ακροατήριο. Μιλούμε για επιστροφή στο μεσαίωνα ουσιαστικά. Ε, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Χίλντε Βάουτμανς από το Άλτε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε με κατάπληξη έμαθα τα νέα και είδα όλες αυτές τις εικόνες από την Τσετσενία. Όταν κανείς βλέπει αυτά τα πράγματα και ακούει αυτές τις μαρτυρίες, νομίζει ότι ε, έχουμε επιστρέψει στο Μεσαίωνα να κρατούνται σε στρατόπεδα κράτησης ομοφιλόφιλοι άνδρες και άνθρωποι για τους οποίους υπάρχει υποψία υποτίθεται ότι είναι ομοφιλόφιλοι και να τους απειλούν τα μέλη της δικής τους οικογένειας και όλα αυτά να συμβαίνουν στη γειτονιά μας στην πίσω αυλή μας εμάς εδώ στην Ευρώπη Έχουμε τη Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας και δεν νομίζω ότι έχουμε λόγους να τη γιορτάσουμε. Αντιθέτως, πρέπει να αυξήσουμε την πίεση που ασκούμε. Αντιθέτως, πρέπει να δράσουμε, να αναλάβουμε δράση, να διασφαλίσουμε ότι τη χάνουν προστασίας οι ομοφιλόφιλοι, να σκεφτούμε τις θεωρήσεις, τις βίζες, τις πρακτικές δικλείδες ασφαλείας και τις εγγυήσει. Όλα αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Άλατ Σμιθ από τους Πράσινους για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που συμφωνούμε όλοι σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Δεν είναι εύκολη δουλειά ε, είμαστε ευγνώμονες στην κοινωνία των πολιτών που μας ε, επέστησαν την προσοχή στο μεγάλο αυτό πρόβλημα η Διεθνής Αμνηστία, το Human Rights Watch και άλλες διεθνείς οργανώσεις ε, κάνουν τεράστιες προσπάθειες και επιδεικνύουν και γενναιότητα. Το θέμα της Τσετσενίας είναι αντικείμενο αυτού του ψηφίσματος, αλλά το πρόβλημα δεν περιορίζεται εκεί. Υπάρχει μια τάση στην πολιτική να δημιουργούνται από δύο πομπέοι, τράγοι ε, και η πρόοδος ε, είναι αναστρέψιμη. Υπάρχουν μεγάλες ισχυρές δυνάμεις που επιτυγχάνουν πολλές φορές να υπονομεύσουν και να παραμορφώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, των μειονοτήτων στον ευρύτερο κόσμο. Έχουμε μεγάλη δουλειά να κάνουμε και ε, μεγάλη δουλειά μας αναλογεί και μας. Υιοθετώ πλήρως το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Γιώζεφ ε, Βάιντεν Χόλτσερ. Ευχαριστώ. Η κατάσταση στην Τσετσενία είναι ανησυχητική εδώ και πολλά χρόνια. Πιο πολύ από ε, άλλες περιοχές στην Ρωσική Ομοσπονδία. Εδώ τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεχώς προκλητικά και συστηματικά παραβιάζονται. Ε, βλέπουμε ότι και δυνάμεις, ε, οι δυνάμεις ασφαλείας συμμετέχουν ή είναι παρατηρητές των ε, βιαιοτήτων κατά των ομοφιλοφίλων. Αυτό σοκάρει. Ε, είναι λογικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και βεβαίως υπάρχει και σαφής θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι οι ε, βιότητες ε, κατά τον ε, ΛΟΑΔΜ κλιμακώνονται κάθετα. Η Ρωσική Ομοσπονδία υπεσχέθη να φωτίσει το θέμα, αλλά αυτά που κάνει δεν επαρκούν επουδενή. Χρειαζόμαστε πραγματικές γνήσιες εξηγήσει. Ευχαριστούμε κύριε Βάιντεν Χόλτσερ. Και τώρα η κυρία Καρίμα Μαντέλη. Ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, Αύριο γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας και την ίδια στιγμή στη Τσετσενία ε, διώκονται οι ομοφιλόφιλοι. Αν είσαι ομοφιλόφιλος εκεί είτε θα βρεις το θάνατο είτε θα πρέπει να πας εξορία. Είναι απαράδεκτο να παραμείνουμε βουβοί μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, μπροστά σε αυτούς που καταστρατηγούν τις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε η φωνή των θυμάτων των διώξεων. Απευθύνουμε έκκληση για την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων απευθύνουμε έκκληση για σοβαρή έρευνα από τους διεθνείς οργανισμούς για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει θάρρος μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στη Τσετσενία, μια χώρα που είναι μέλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας του κυρίου Πούτιν. Η ίδια Ομοσπονδία θα υποδεχθεί ε, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, κάποιοι θα παίζουν ποδόσφαιρο και άλλοι θα σφαγιάζονται όσο τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν τηρούνται στη Ρωσία και στις δορυφόρους της, ε, σας καλώ να ε, απόσχουμε από οποιοδήποτε είδους ε, τέτοια δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σιλβί Γκυγιόμ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Το 2013 το επιθυμήσατε κι εσείς κύριε Επίτροπε, χαιρετήσαμε την υιοθέτηση από το Συμβούλιο των Κατευθυντήριων Γραμμών για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ και θεωρήσαμε ότι έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να καταπολεμήσουμε την ομοφοβία. Ωστόσο, τέσσερα χρόνια αργότερα ε, παραμένουν, οι, τα, παραμένουν θύματα διακρίσεων και βίας τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ένας νόμος ομοφοβικός ψηφίστηκε στη Ρωσία πριν από τέσσερα χρόνια και ε, αυτό το δηλητηριώδες ε, κλίμα έχει οξυνθεί. Ε, γίνεται ουσιαστικά δεν, δέχονται τη διαφορά, το διαφορετικό των άλλων και έχουμε, έχουν καταντήσει να υπάρχουν πραγματικά τερατώδεις καταστάσεις. Αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι η ανθρώπινη ζωή. Θα πρέπει να δώσουμε ένα ασφαλές καταφύγιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι Ευρωπαίοι πρέσβεις θα πρέπει να τους δώσουν βίζα για να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ρωσικές αρχές θα πρέπει να ρίξουν άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση και να σεβαστούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τερένε Ράιντκε, παρακαλώ, από τους Πρασίνους. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι, αυτά που συμβαίνουν στην Τσετσενία σήμερα είναι η πιο ακραία κλιμάκωση της επίθεσης εις βάρος των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ διώξεις, ακόμα και δολοφονίες. Ε, είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Προϋπόθεση όμως από αυτές τις απάνθρωπες ενέργειες είναι η άρνηση του ότι υπάρχουμε. Οι ομοφιλόφιλοι άνδρες, γυναίκες, τρανς, μπάι, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αρνούμεθα ότι υπάρχουν. και όμως το καθεστώς στη Ρωσία αρνείται την ύπαρξή μας και γι' αυτό δεν μπορούμε απλά να μην κάνουμε τίποτα, να μείνουμε αδρανείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει και να προασπιστεί τα δικαιώματα αυτών των οποίων η ίδια η ύπαρξη δεν αναγνωρίζεται. Τότε θα είμαστε υπερήφανοι που υπάρχουμε. Ευχαριστώ Βιώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, μπορεί κανείς ε, να αντισταθεί σε επιθέσεις οι οποίες γίνονται με πραγματικά όπλα, αλλά Πραγματικά ο πόνος τον οποίο έχει νιώσει κανείς με τέτοιου είδους καταστάσεις μετά από βασανιστήρια και αυτά μας τα λέει ο Αντρέη ο οποίος βασανίστηκε όπως και εκατοντάδες άλλοι στην Τσετσενία. Πραγματικά είναι το καθεστώς φρίκης του Καντήροφ τον οποίο προστατεύει ο Πούτιν και θυμίζω ότι στη Μόσχα συνελήφθησαν τρεις υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ μεταξύ και των οποίων ένας Ιταλός. Είναι κόλαση η ζωή στην Τσετσενία, ιδιαίτερα για τους ομοφιλόφιλους. Συλλαμβάνονται, βασανίζονται, κρατούνται ε, και πολλές φορές ε, οθούνται οι οικογένειες σε εγκλήματα τιμής. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να εκφράσει την αγανάκτησή της για την κατάσταση αυτή. Τι είναι η Ευρώπη αν δεν διασφαλίσει και υπερασπιστεί ε, όλους αυτούς των οποίων η ίδια η ζωή είναι σε κίνδυνο. Θα πρέπει η Ευρώπη λοιπόν σήμερα ε, να μην αποστρέψει την κεφαλή και να ε, κοιτάξει κατάματα τους Ρώσους και να τους ζητήσει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Με τις χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θέλουμε καμία επαφή. Δεν μπορούμε να αντέχουμε τις παραβιάσεις εις βάρος των θρησκευτικών δικαιωμάτων, τις παραβιάσεις εις βάρος των δικαιωμάτων των γυναικών, των ομοφιλοφίλων. Όλα αυτά είναι επιθέσεις στις αξίες της Ευρώπης και απαιτείται μια αυστηρή απάντηση. Ευχαριστώ τον κύριο Βιώτη. Ντάνς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς τον Επίτροπο που μας εξήγησε την προσπάθεια που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς το συζητάμε το θέμα αυτό λόγω της σκληρής δουλειάς που έκανε η κοινωνία των πολιτών. Εμείς ε, ε, οι αντιδράσεις της Ρωσίας και της Τσετσενίας, οι οποίες αρνούνται την ύπαρξη του προβλήματος, ε, μας απογοητεύουν. Και δεν μπορούμε παρά να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς των οποίων η ζωή απειλείται. Εγώ ίδιος είμαι γκέι και μαζί με τους υπόλοιπους ΛΟΑΔΜΑ Θέλουμε να εξηγήσουμε το τι κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να με συλλάβουν, Εγώ μενα δεν θα με συλλάβουν οι αρχές, δεν θα με πετάξουν στον δρόμο μετά από τον ξυλοδαρμό μου. Γιατί η κυβέρνησή μου και η κοινωνία με προστατεύει. πρέπει να κατανοήσει κανείς ότι το πρόβλημα δεν είναι οι ομοφιλόφιλοι, το πρόβλημα είναι αυτοί που διώκουν τους ομοφιλόφιλους και γι' αυτό η διεθνής κοινότητα πρέπει να τους υπερασπιστεί. Σας ευχαριστώ κύριε Ντάνς για μια εντυπωσιακή παρουσίαση λέει ο πρόεδρος η κυρία Ward. Ένα λεπτό. Ποτέ δεν θα επιτρέψουμε την τυρονία της πλειοψηφίας να καταπιέζει την μειοψηφία έλεγε ο κύριος Κάσμαν στα πλαίσια των Ολυμπιακών του 2014 στο Σότσι. Μετά από τρία χρόνια βλέπουμε ότι δεν μπορούμε εμείς να ανεχόμαστε αυτές τις συμπεριφορές. Οι διώξεις των ομοφιλοφίλων και των φερόμενων ως ομοφιλοφίλων είναι απαράδεκτες και πρέπει να τερματιστούν. Ο κύριος Πούτιν είπε ότι θα υποστηρίξει μια ερεύνηση της υπόθεσης μετά από πίεση ε, της κυρίας Μέρκελ. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει την πίεση εις βάρος των Ρώσων. Ο Ιταλός εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήθελε να καταθέσει μία αναφορά με δύο εκατομμύρια υπογραφών για τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων στη Ρωσία συνελήφθη μεν αλλά απελευθερώθηκε μετά από λίγες μέρες λόγω της πίεσης της κοινή γνώμης. Πρέπει να υπερασπιστούμε αυτούς που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτών οι οποίοι πολεμούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό τους. Κλάβδιαν Φροντσούλιτσα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία όλο και πιο ανησυχητική γίνεται. Εκατό χιλιάδες άνθρωποι στην Τσενία και στη Ρωσία έχουν συλληφθεί, κατηγορηθεί για ομοφιλοφιλία, έχουν ε, βασανιστεί ε, στις φυλακές, ε, υπήρξε και ένας θάνατος στη φυλακή, αντιμετωπίστηκαν απάνθρωπα κάτω από φρικτές συνθήκες. Οι αρχές αρνούνται τις κατηγορίες αυτές και λέγουν ότι δεν ε, υπάρχουν φερόμενοι ως ομοφιλόφιλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση. Θα πρέπει να ενημερωθούμε για τα μέτρα που έχουν συγκεκριμένα ληφθεί και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές ώστε να προστατεύονται ε, οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρκ Ταραμπέλα, παρακαλώ. δεν ρωτώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η ελευθερία να είναι κανείς ομοφιλόφιλος είναι δικαίωμα, αλλά όχι στη Τσετσενία, όπου ο Πρόεδρος αποφάσισε να εξολοθρεύσει όλους τους ομοφιλόφιλους μέχρι τις 26 Μαΐου αξιόπιστες πηγές δείχνουν ότι υπάρχει ένα στρατόπεδο κράτησης, ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου δεκάδες γκέι αποθηκεύονται εκεί, συσσωρεύονται, βασανίζονται και ενδεχομένως σκοτώνονται. Ε, καλούνται οι οικογένειες να σκοτώσουν τα ομοφυλόφιλα παιδιά τους ε, για να ξεπλύνουν την τιμή της οικογένειάς τους μιλούμε για ε, καθάρσεις ολόκληρες πληθυσμών, ε, αιμοσταγής Είναι μια απάντηση εμετική ουσιαστικά αυτή που επιφυλάσσει το καθεστώς στην κοινότητα αυτή των ανθρώπων. Οι ευρωπαϊκές μας αξίες μας απαγορεύουν να παραμείνουμε βουβοί και αμήλυτοι και τυφλοί. Προτείνουμε επιγόντως να δοθεί βίζα ε, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στις πράξεις και να μην μείνουμε στα λόγια. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταραπέλα, λέει ο Πρόεδρος. Προχωρούμε στη διαδικασία Catch the Ο κύριος πώς είναι ο πρώτος ομιλητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μίλησαν εδώ. Είναι καθαρή η φωνή μας που καταδικάζει την κατάσταση στην Τσετσενία, που καταδικάζει την μοίρα των ομοφιλοφίλων που αντιμετωπίζουν διακριτική μεταχείριση, απειλούνται και απειλείται και η ζωή τους. Ε, χαίρομαι που και ο Επίτροπος αναφέρθηκε στα ζητήματα αυτά. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στην αντιμετώπιση μας. Είμαι και επιφυλακτικός. Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν έχει υπόψη του να κάνει κάτι μια σε βάθος ανάλυση για να αναδείξει το τι συνέβη στην Τσετσενία. Οι άνθρωποι που διώκονται νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσουν βίζα και να πάρουν και άσυλο και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα ανεξάρτητα, τις ανεξάρτητες οργανώσεις που τα αποκαλύπτουν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Τα νέα που έρχονται από την Τσετσενία και τη Ρωσία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Συστηματικά βασανιστήρια, κρατήσεις ε, ε, εκατοντάδων ομοφιλοφίλων ή φερόμενων ως ομοφιλοφίλων, όπως επίσης και στρατόπεδα αναμόρφωσης ε, και φυλάκισης, σκοτεινές σελίδες της ανθρωπότητας και η σύλληψη των τελευταίων, τελευταία των ακτιβιστών στη Μόσχα, μεταξύ των οποίων και ενός Ιταλού, δείχνει ότι πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε τις πιέσεις αυτές. Πρέπει να πιέσουμε αντίθετα τις ρωσικές αρχές για να αλλάξουν ε, πρακτική. Αύριο είναι η Διεθνής ημέρα για την ομοφοβία και θα πρέπει να πούμε ότι και στην Ιταλία στα πλαίσια του ε, Pride της Reggio, στο Reggio Emilia θα πρέπει να αναγνωρίσουμε για μια ακόμη φορά ε, την ελευθερία του καθενός να συμπεριφέρεται στην ερωτική του ζωή όπως αυτός επιλέγει. Ευχαριστώ. Gracias, ο νόμος του 2013 εις βάρος των νομοφιλοφίλων στην Ρωσία επέτρεψε στο καθεστώς Καντήροφ να κάνει αυτά τα οποία κάνει σήμερα. Είναι τεράστιος ο αριθμός βέβαια των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρωσία. Και με ευκαιρία την ημέρα εναντίον της ομοφοβίας θα ζητήσω να βοηθήσουμε την προσφυγή και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τις ενέργειες του καθεστώτος εις βάρος των ομοφιλοφίλων. Όσο ισχυροί και αν είναι θα πρέπει να τους παραπέμψουμε στη διεθνή δικαιοσύνη. Εμείς θα ζητήσουμε ε, την αποποινικοποίηση ε, στα πλαίσια των εκδηλώσεών μας της ομοφιλοφιλίας σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Καστάλντο έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση η οποία ισχύει στην Τσετσενία είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Και οι καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν στην ΟΒΑ για Γκαζέτα δείχνουν απαράδεκτες συνθήκες για την σύλληψη, κράτηση, βασανισμό και εξύβριση των ομοφιλοφίλων, όπως επίσης και πιέσεις προς τις οικογένειες για εγκλήματα τιμής εις βάρος των ομοφιλοφίλων ε, λέγοντας ότι ο οικογενειακός ιστός ε, κινδυνεύει λόγω των ανθρώπων αυτών. Νομίζω ότι οι ενέργειες του Καντήροφ και της Σαράτοβα ε, είναι απαράδεκτες και πράγματι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Εμείς ζητάμε να γίνει κάθε προσπάθεια από πλευρά των ρωσικών αρχών για να αλλάξει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση και να προστατευθούν τα θύματα όπως και οι οικογένειές τους. Αυτό νομίζω είναι το ελάχιστο το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Καστάλντο. Εξ τώρα λοιπόν της ε, κυρίας Μογκερίνη, ο κύριος Τηλιανίδης έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ που δείχνετε αυτήν την ενότητα στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Όλοι συμμεριζόμεθα την ανησυχία για τα τεκτενόμενα στην Τσετσενία. Όλοι συμφωνούμε ότι το ζήτημα αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και πιστεύω προσωπικά ότι είναι ντροπή να πρέπει να συζητάμε το, ένα τέτοιο ζήτημα σήμερα τον 21ο αιώνα. Η βία σε βάρος της κοινότητας των ΛΟΑΔΜΑ ε, ε, ανέδειξε την ε, πολύ αρνητική κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτήν την Ρωσική Ομοσπονδία. Θα συνεργαστούμε για να στηρίξουμε τα θύματα και θα πιέσουμε τις ρωσικές αρχές για να σταματήσει την βία και να εξασφαλίσει δικαιοσύνη για τα θύματα. Παρακαλώ να γνωρίζετε ότι κάποιες κοινέ μας προσπάθειες θα απαιτήσουν α, υπομονή και εμπιστευτικότητα. Όλοι προσπαθούμε να βοηθήσουμε βεβαίως, αλλά και μπορούμε να κοινοποιούμε τις ε, προσπάθειές μας. Όμως καμιά φορά είμαστε πιο, είναι πιο σημαντικό να είμαστε αποτελεσματικοί παρά ε, ε απόλυτα ειλικρινοί στις δηλώσεις μας. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί γνωρίζω κάποιες περιπτώσεις επιτόπου. Θα ήθελα να κλείσω τονίζοντας άλλη μια φορά την εκτίμησή μου για τον ρόλο του Κοινοβουλίου που διατήρησε στην ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό. Πρέπει να συνεχιστεί η πάλι για να δείξουμε την προθυμία μας, την ισχυρή μας πεποίθηση σχετικά με τα δικαιώματα της κοινότητας των ΛΟΑΔΜΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ιδιαίτερα για όσα είπατε σχετικά με το καθήκον και το ρόλο μας, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κλείνουμε λοιπόν την συζήτηση. Έχω ε, λάβει έξι σχέδια ψηφισμάτων από τις έξι μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες. Η ψηφοφορία θα